στις φορολογικές και άλλες και τα εργασιακά δικαιώματα όπως επίσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Ζωρίνιο έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει ότι είναι γεωπολιτική πολιτική και την ενδιαφέρουν οι σχέσεις με την Αφρική έτσι το αποδεικνύει αυτό. Στο γεωπολιτικό λοιπόν πλαίσιο η Αφρική εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια και πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε εταιρικέ σχέσεις στρατηγικής σημασίας. Αυτή η στρατηγική σχέση με την Αφρική ανταποκρίνεται στα ε, συμφέροντα των λαών και πρέπει να είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τα λάβουμε υπόψη μα σε κάθε διάσταση. Συνεπώς, πρέπει να στοιχηματίσουμε υπέρ τη κοινωνία των πολιτών, να διασφαλίσουμε τη συνοχή και την σαφή διάρθρωση της πολιτικής αυτής με την συμφωνία μετά το Κοτονού, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες. Και επίσης να συμμετέχουν τα κοινοβούλια, να υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση, δηλαδή στην εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ και στις σχέσεις του Κοινοβουλίου μας με το Αφρικανικό Κοινοβούλιο. Έτσι θα πετύχουμε μαζί. Ευχαριστούμε. Επόμενος, η κυρία Ζαχαροπούλου έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ, για 1,5 λεπτό. Madame la commissaire, chers collègues. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ας δούμε την Αφρική το 2020. Έχει ένα νέο πρόσωπο της νεολαίας της, των γυναικών της. Η Αφρική είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ε, με επιτυχία. Και ό,τι κάνει σήμερα θα έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον του κόσμου. Α δούμε τώρα την Ευρώπη το 2020, μια ήπειρο αξιών, εμπειριών, που είναι όμω ταυτόχρονα μια ήπειρο πόλο και περισσότερο, που πιο πολύ από ποτέ έχει ανάγκη από συμμάχου. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή περήφανη Αφρική, Όπω και η Αφρική χρειάζεται μια ενωμένη Ευρώπη που θα μιλάμε μια ενιαία φωνή. Και αυτή είναι η προπόθεση ώστε το πολυμερέ σύστημα να επιβιώσει και να επιτευχθούν οι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κυρία Επίτροπη, είναι στρατηγική. Θα πρέπει να ενσαρκώσει μια νέα νέα σχέση ανανεωμένη μεταξύ των δύο υπήρων. Θα πρέπει να τεθεί οριστικό τέρμα στη μεταπικιοκρατική εποχή και στα σχετικά αφηγήματα γιατί οι Αφρικανοί ε, σύμμαχοί μας ζητούν μια ισότιμη σχέση. Αλλά και εμείς Ευρωπαίοι θέλουμε να γράψουμε μια νέα σελίδα μαζί με τους Αφρικανούς. Μια νέα στρατηγική όχι για την Αφρική αλλά μαζί με την Αφρική. Και έχουμε και ένα άλλο καθήκον. Το χρέο να επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους να καταλάβουν, να κατανοήσουν την Αφρική υπό όλο το φάσμα και όλες τις πτυχές όχι μόνο αυτή τη μετανάστευση. Το νέο σα χαρτοφλάκ περιλαμβάνει τη λέξη διεθνεί τερικέ σχέσει. Και αυτό ανοίγει νέα σελίδα στην ιστορία μα. Ω βουλευτή είμαι περήφανη που μπορώ να συγγράψω αυτό το κεφάλαιο μαζί σα με τι συμβουλέ, με του συναδέλφου μου και με του συμμάχου μα από την Αφρική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Αλένα για ένα, Για ένα λεπτό. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, μετά το τέλο τη απικιακή εποχή και τη ανεξαρτησία των κρατών τη Αφρική, η Ένωση πολλαπλασίασε τι συμφωνίε συνεργασία με την Αφρική. Σίγουρα είχαμε τι συμφωνίε του Γιαουντέ, του Λομέ, τη συμφωνία του Κοτονού και πολλέ άλλε. Αλλά οι περισσότερε αυτέ συμφωνίε Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι σίγουρα καθόριζαν τι δικέ μα σχέσει με την Αφρική, αλλά πολύ συχνά ήταν εκεί για να διατηρήσουν την επιρροή μα και τα συμφέροντά μα επί τη Υπήρου. Ο απολογισμό μετά από μισό αιώνα συνεργασία δεν είναι λαμπρό, δεν είναι λαμπρό αν δούμε του δείκτε του αναπτυξιακού, αν δούμε την ποικιλομορφία την οικονομική, αν δούμε τι ανισότητε ή ακόμα τα θέματα τη ασφαλεία όσον αφορά την Αφρικανική Ήπειρο. Λοιπόν, δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τι σχέσει μα από την Αφρική και χαιρετίζω την πρωτοβουλία για τη μελλοντική στρατηγική Ευρωπαϊκή Ενώσεω Αφρική. Αλλά εξυπακούεται ότι θα πρέπει να αποδείξουμε περισσότερη συνοχή και να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Η συνοχή μεταξύ των διαφόρων μέσων που χρησιμοποιούμε και αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια των ε, στόχων της Ε, θα πρέπει να έχουμε συνοχή όσον αφορά τι πολιτικέ μα. Δεν μπορούμε, παραδείγματο χάρη, να Έχουμε μια εμπορική συμφωνία που δεν ευνοεί την περιφερειακή ανάπτυξη και που καταστρέφει ε, την τοπική γεωργία προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών. Θα πρέπει επίσης να επικρατεί διαφάνεια και να υπάρχει και χρηστή διακυβέρνηση. Ναι λοιπόν για μια στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, αλλά μην ξανακάνουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος πάει στην κυρία Ροντρίγκες Ράμους για ένα λεπτό. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις στο ΚΑΣΤΙΑΕ. Παρακαλώ να έχουν όλοι το χρόνο να μιλήσουν. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο που σας διατίθεται. Ευχαριστώ. το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Η Αφρικανική Ήπειρος δεν είναι ήπειρος μόνο της μετανάστευσης αλλά και του μέλλοντος, των νέων και των γυναικών που όλο και περισσότερη δύναμη έχουν και μπορούν και πηγαίνουν όλο και πιο μακριά. Αυτή λοιπόν η νέα στρατηγική της Ευρώπης θα πρέπει να είναι μια πράσινη στρατηγική, πολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθαρές ε, ενέργειες. Αυτά πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της νέας μας σχέσης με την Αφρικανική Ήπειρο. Τον τελευταίο αιώνα η Αφρική συνεσέφερε με 2% μόνο ε, εκπομπές ε, στην θέρμανση του πλανήτη. Όμως υφίσταται τι χειρότερε συνέπειε γιατί η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα και είναι ακριβώ στην Αφρική όπου πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι εξαιτία τη ξηρασία Η ε απο τι πλημμύρε. οποτε χρειάζεται περισσότερους πόρους, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα αυτό χρειαζόμαστε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πισαρία. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στη σημερινή συζήτηση μια μόνα λέξη επαναλήφθηκε τις περισσότερες φορές. Η λέξη μετανάστευση. Γνωρίζοντα τη σημαντική πόσο σημαντική είναι και τις προκλήσει που δημιουργεί, είμαι ότι η ανάπτυξη η κοινωνική, η οικονομική και η δημοκρατική είναι και θα πρέπει να είναι ο στόχος που έχει προτεραιότητα. Ε, θέλουμε, για να θέσουμε τροχοπέδι στη μετανάστευση πρέπει να, έχουμε, ε, να σταματήσουμε την αναποτελεσματική αδύναμη ε, πολιτική μας. Η ειρήνη και η ανάπτυξη είναι το DNA της Ευρώπης. Πρέπει να τη μοιραστούμε με το λαό της Αφρικής και να σταματήσουμε τα λάθη του παρθόντος. Τα ευρωπαϊκά χρήματα πρέπει να δίνονται για την ανάπτυξη της Υπήρου και όχι να χρηματοδοτήσουν ε, διάφορα έργα που δεν συμφωνούν με του στόχου μα. Το 2020 θα έπρεπε να είναι η χρονιά τη καμπή όσον αφορά τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Κλείνω με αυτά που είπε ο Νέλσον Μαντέλα. Κανεί δεν γεννήθηκε σκλάβο, ούτε κύριο, ούτε για να ζει στη μιζέρια. Αλλά όλοι γεννηθήκαμε για να είμαστε αδέλφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ραφαέλα για ένα λεπτό. Κυρία επιτροπή, κυρία... συνάδελφοι, ευχαριστώ την πρόεδρο, την κυρία Βαντελάιν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έκανε το πρώτο διεθνέ ταξίδι στην Αφρικανική Ένωση. Είναι σημαντικό μήνυμα. Η Αφρική και η Ευρώπη είναι σαν σταυροδρόμι και θα πρέπει να αλλάξουμε την όλη νοοτροπία μα. Είναι και η ώρα να θεωρήσουμε ε, ότι είμαστε ίσοι και έχουμε αυτή την Ήπειρο που είναι στην πόρτα μα και μπορούμε να λάβουμε πρωτοβουλίε που υπόσχονται πολλά. Η Αφρικανική Ήπειρο μπορεί να έχει μια ζώνη ελευθέρου συναλλαγών. Είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα φιλόδοξο έργο που μπορεί να μεταμορφώσει την Αφρική και να γίνει ε, πολυμερής ε, περιοχή για το εμπόριο. Α κάνει ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη δημιουργία Τη ε, ζώνη για ελεύθερο εμπόριο στην, Αφρικανική, στην Αφρικανική Ήπειρο. Θα πρέπει αυτό να αντικατοπτρίζεται και στο σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένα μέτρα και είναι προ το δικό μας όφελος να έχουμε μια ενωμένη Αφρικανική Ένωση. Πρέπει να το εστερνιστούμε αυτό. Άλλοι προσπαθούν να ενωθούν όταν σήμερα υπάρχουν κάποιε. Ε, δυνάμεις που κινούνται εναντίον μα. Και η σύμπραξη μεταξύ Αφρικανικών χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι μια ένωση μεταξύ ε, ομοτήμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλούς συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Δεν θα έχουν όλη τη δυνατότητα να μιλήσουν όμω. Πρώτο, στον κατάλογο ο ω Μίλαν Μον. Παρακαλώ να θυμηθείτε ότι έχετε ένα λεπτό καθένας. Ευχαριστώ. Η Αφρικανική Ήπειρο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Πρέπει να συνεισφέρουμε στην ειρήνη, στην ασφάλεια, στην ανάπτυξή τη, αλλά και στους θεσμούς τη και στην ολέα τη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι μεταναστευτικέ ροέ από την Αφρική να έρχονται συντεταγμένα. Είναι μια ήπειρο με τεράστια δημογραφική ανάπτυξη. Τη χρειαζόμαστε την Αφρική και η διάσκεψη κορυφή του επόμενου εξαμήνου θα είναι πολύ σημαντική. Θέλω τώρα να αναφερθώ στο, στην ε, πιο γειτονική μας Αφρικανική Ήπειρο. Είχαμε τη διαδικασία της Βαρκελόνης. Δεν καταφέραμε όμως να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο ευημερία, σταθερότητας και ελευθερίας που θέλαμε στη Βόρεια Αφρική. Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχώρησε. Τι ξένες δυνάμεις υπάρχουν στη Συρία, ποιος πρωταγωνιστεί στη Λιβύη, ποιος ε, τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά στην ευτική διαδικασία στην, ε, ε, ε στην Ανατολή. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά, αλλά και βέβαια επιρροή στην Αφρική και στην ε, νότια πλευρά της Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκε Μάρκες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως και εδώ έτσι και εκεί δημιουργούν περιέργεια και προσφέρουν και ευκαιρίες. Ευκαιρίες για νέες λύσεις σε διάφορα προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων με μία εφαρμογή όπως μας το έδειξαν εδώ κάποιοι νέοι από την Κένια μπορεί να γίνει. Επιτέχουμε τα εικονικά νομίσματα. Έχουμε... Είδαμε τι έχει γίνει στην Μοζαβίκη και αλλού. Η τεχνολογία λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί στην Κάνα και αλλού για τα ψηφιακά. Η ανάπτυξη αυτή της τεχνολογίας φέρνει βέβαια και κινδύνους. Χρειάζεται λοιπόν κατάρτιση, χρειάζεται οι γυναίκες, οι νέοι να μαθαίνουν. Αυτά είναι στοιχεία εξίσου σημαντικά για την Αφρική όπως είναι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς η στρατηγική αυτή θα πρέπει να προωθήσει και να κάνει πιο στενές τις σχέσεις μας, την εταιρική μας σχέση με την Αφρική, που πρέπει να βλέπουμε σαν έναν εταίρο με ευκαιρίες και προκλήσεις όπως έχουμε και εμείς εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κέμπα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε θερμά για την νέα αυτή προσέγγιση και για τη νέα στρατηγική για την Αφρική. Είναι κάτι πραγματικά αναγκαίο, το συζητήσαμε και στην Επιτροπή ΝΤΕΒΗ και σας ευχαριστώ για την ε, στάση σας. Έχουμε πολλές μεταξύ των διαφόρων φυλών, ανεργία, έλλειψη απασχόλησης για τους νέους. Και όλα αυτά είναι πρόβλημα ε, και οδηγεί στη λαφρομετανάστευση, αλλά είναι και ένα φαινόμενο το οποίο εξυκολουθούμε να παρατηρούμε στην Αφρική, η εμπορία ανθρώπων. Ε, και στην Πολωνία ξεκινήσαμε μία μείζωνα δράση. Συλλέγουμε δωρεές μέσω δύο οργανώσεων για να υποστηρίξουμε αυτούς ή αυτές που κατάφεραν να γλιτώσουν από την πρακτική αυτή. Και γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε παιδιά, γιατί πολλούνται, ε, ε, μέχρι και πεντάχρονα κορίτσια ε, πολλούνται και χρησιμοποιούνται, τις εκμεταλλεύονται ως πόρνες. 300 δολάρια κοστίζει ένα αγόρι, ε, για να σας ένα παράδειγμα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, πρέπει να συμπεριλάβουμε το θέμα στην είναι αυτή η στρατηγική. Δεν μπορούμε ε, να επιτρέψουμε να γίνεται νόμιμα η σωματεμπορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Είναι σημαντικότατο να θεωρήσουμε ότι η Αφρική είναι ισότιμος εταίρος σε αυτή τη νέα στρατηγική. Πρέπει να έχουμε μια πραγματική ε, συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της του κλίματος και άλλα θέματα. Στην Αφρική, η ανάπτυξη της Αφρικής είναι κρισίμου σημασίας και έχει σημασία για όλο τον κόσμο. Είναι μια τεράστια ήπειρος ε, η Αφρική. Επίσης, αυτό που είπε και ο Τόμπε είναι σημαντικό, ότι αν θέλουμε να συζητήσουμε τα πάντα που ανέφερε και ο Τόμπε, θα χρειαζόμαστε μια εβδομάδα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μόνο ένα πράγμα, το ρόλο ε, των γυναικών και των κοριτσιών και ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των γυναικών που μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ζωής όλων. Καμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρί να λαμβάνει υπόψη το 50% του πληθυσμού τη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κορίτσια θα μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, ότι θα έχουν δικαίωμα να έχουν σεξουαλική υγεία και τα παιδιά ή τα κορίτσια θα πρέπει να παντρεύονται θελοντικά και όχι καταναγκαστικά και ελπίζω όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει η Ντέρτρι Κλούν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, επρόσδεκτη η κλουν ευχαριστω κυρια προεδρε επιτροπε επροσδεκτη δηλωση σας που είπατε ότι πήγατε με την κυρία Βοντελάιν στην Αφρική για να ακούσετε τη φωνή της Αφρικής. Σημαντική, πολύ σημαντική ε, κίνηση αυτή. Είναι γεμάτη δυναμικότητα με τους νέους της Αφρική. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη συνεργασία μας, ε, τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Αφρικής. Είναι καλή στιγμή. Νομίζω ότι είχαμε επιτυχίες, αλλά τώρα έχουμε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε τη Συμφωνία για την Αλλαγή του Κλίματος των Παρισίων και πρέπει να ανανεώσουμε ε, την προσοχή που θα δώσουμε στη σχέση μας αυτή. Ιδιαίτερα πιστεύω ότι, ότι τα θέματα που άπτονται της ανεργίας, που είναι σε ψηλά επίπεδα, ε, μπορεί να, η καταπολέμηση της ανεργίας μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη θέσεων. Εγώ επισκέφθηκα επανειλημμένα την Αφρική στην προηγούμενη θητεία και είδα ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει η Ευρώπη υποστηρίζοντας ε, την ντόπια βιομηχανία για να αναπτύξουν θέσεις απασχόλησης και να βοηθήσουμε και με την ανάπτυξη της παιδείας. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να αναπτύξουμε μια νέα στρατηγική, ανανεωμένη στρατηγική με τους γείτονές μας στην Αφρική. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Αφρική μπορεί να συνοψιστεί χαλαρά ως εξής. Πολύ γλυκά λόγια, που λέμε στο Κοινοβούλιο, μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ισότητα, αλλά ποικιλοτρόπος απλώς είναι φίλος για την, για την παγκοσμιοποίηση την οφειλελεύθερη και τα βλέπουμε σε πολλές διευθετήσεις εμπορικές όπου λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ΑΚΕ χάνουν τις εξαιρέσεις δασμών ε, σε αμοιβέ σχέσεις ενώ η γεωργία ευρωπαϊκή κρατά προστατευτικούς μηχανισμούς που έχουμε υιοθετήσει εμείς για την ε, περιοχή μας. Οι νεοφιλελεύθερες εμπορικές συμφωνίες είναι το μόνο χαρακτηριστικό ανισόρροπης σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης και Αφρικής. Ιδιαίτερα πρέπει να προβληματιζόμαστε για να αυξανόμενη στατιωτική παρουσία, κυρίως στο Σαχέλ, κυρίως από τους Γάλλους, που βοηθούν δικτάτορες στην περιοχή, ούτω ώστε να υποστηρίξουν τα γαλλικά συμφέροντα για πρώτε ύλε και φθηνά εργατικά χέρια. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να πούμε ότι είναι ισότητα, δεν κάνει καλό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τελευταίος ομιλητής, Κρίστοφ Χέτμαν. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα στρατηγική για την Αφρική πρέπει να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ε, συνθήκες ε, και στην πραγματικότητα. Βάσει οποιασδήποτε συμφωνία, οποιονδήποτε σχέσεων θα πρέπει να είναι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προωθηθεί η ελευθερία λόγου, να εισαχθούν δημοκρατικά πρότυπα. Και για να πετύχουμε αυτό το στόχο θα πρέπει να βαθύνουμε τον πολιτικό διάλογο και από την Αφρικανική Ένωση να εστιάσουμε στην ειρήνη, την ασφάλεια, τον περιορισμό τη φτώχεια τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματο, του συστήματο υγεία, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και την εμπορία ανθρώπων. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να δώσουμε στι χώρε που παλεύουν με αυτά τα σοβαρά προβλήματα, να δώσουμε οικονομική βοήθεια. Έχουμε και την κλιματική δράση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τι πρωτοβουλίε τη Αφρικανική Υπήρου για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ουρπιλάινεν για να μας κάνει την καταλητική της δήλωση. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε. Πρέπει να σας πω πως εγώ έχω εμπιστοσύνη στην δυνατότητά μας να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική και εταιρική σχέση με την Αφρική που επικεντρώνεται στην βιώσιμη ανάπτυξη. Η δικιά σα συνεισφορά στη στρατηγική αυτή είναι στοιχείο κλειδί στη διαδικασία για να διαμορφώσει τη βάση της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, σχεδιάζουν τώρα και συντάσσουν τη στρατηγική αυτή ώστε να είναι γίνεται περισσότερο συνολική. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. σας παρακαλώ να είσαστε σίγουροι ότι τα σχόλιά σας εδώ που έγιναν σήμερα τα σημειώσαμε και χαίρομαι πολύ που ήταν τόσοι πολλοί από εσά που αναφέρθηκαν στην ολέα, στους νέους. Η στρατηγική μας θα αποτελέσει μια σημαντική αλλαγή και θα ενισχύσει την εταιρική μας σχέση με την Αφρική. Η στρατηγική θέλει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις που από μόνη της η μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και να αγνοήσει. Έτσι λοιπόν μας ενδιαφέρει αυτή η εταιρική σχέση. Δημιουργούμε με τον επικεφαλής διαπραγματευτή για τις χώρες ΑΚΕ, τον Υπουργό Ρόπερ Τουσέ από το Τόγκο και ξέρει ότι θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στα τέλη του Μαρτίου για τη συμφωνία μετά την Κοτονού. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μετά και την διάσκεψη Αφρικανικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα συμμετέχουν όλες οι πλευρές ώστε να μπορέσουμε έτσι να σχεδιάσουμε μαζί τη στρατηγική μας. Θα φροντίσουμε συγχρόνως να διασφαλίσουμε και την υλοποίηση των πολιτικών μας έχοντας καταλήξει όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έγκαιρα. Συνεπώς, αξιότιμοι προβουλευτές, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ε, τις δυνάμεις όλων των θεσμικών μας οργάνων για να προχωρήσουμε. Και μόνο μαζί, πραγματικά μόνο μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ασφαλή, βιώσιμη κοινότητα, ώστε να βοηθήσουμε τον πλανήτη να ξαναβρει την υγεία του και να μπορέσουμε μέσα σε αυτόν να ζήσουμε όλοι καλά τις ζωές μας. Ε, περιμένω και προσβλέπω σε συνέχιση του διαλόγου μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνει εδώ η συζήτηση για το θέμα αυτό. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι δηλώσει του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του μίσους στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι για να συμμετάσχετε στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ ή τη μπλε κάρτα, μπορείτε να ε, το ζητήσετε είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι οδηγίες εξάλλου υπάρχουν στην είσοδο του ημικυκλίου. Η Νικολίνα Μπριάτση τώρα θα μιλήσει εκ μέρου του Συμβουλίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι βουλευτές, Πρόσφατα εορτάσαμε την 25η επέτειο από την Απληφθέρωση στο Άζουβιτς και αυτή η επέτειο από την απελευθέρωση του Auschwitz και αυτή η συζήτηση σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικότερη από ποτέ για πολλά ε, χρόνια. Έχουμε ε, τη ρητορική μίσους, εγκλήματα μίσους, ξενοφοβία ε, και αντισημισμό να αυξάνονται στην Ευρώπη. Οι μειονότητες και άλλες ευάλωτες ομάδες ε, και Εβραίοι πλήττονται και σημειώνουμε το ότι υπάρχει έντονο αντισημιτικό μίσος ακόμη και σήμερα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό το φαινόμενο και είμαστε υποχρεωμένοι αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίζουμε με, με άκρα σοβαρότητα. Υπάρχουν νομικά μέσα τα οποία προσφέρουν προστασία κατά ε, μορφών μυσαλλοδοξίας όπως είναι ο ρατσισμός. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεχθεί τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάρριση οποιασδήποτε μορφής ε, φιλετική διάκρισης. Έχουμε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που απαγορεύει διακρίσεις λόγω φύλου, χρώματος, εθνοτικής ε, καταγωγής, ε, θρησκευτικής πεποίθησης κτλ. Και υπάρχει και ειδική νομοθεσία για την καταπολέμηση της της μυσαλλοδοξίας και του μίσους. Το 2008 ελήφθη μια απόφαση για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Στον Ιούνιο του 2016 το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν αποτελεσματικά ε, στην Εθνική Νομοθεσία τη Συμφωνία Πλαίσιο και άλλη νομοθεσία σχετικά με τη ρητορική μίσου στο Εθνικό Δίκαιο και ζήτησε επίση από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικά μέτρα υποβολή αναφορών, καταγραφή ε, εγκλημάτων μίσου. Στι 6 Δεκεμβρίου το 2018 τα κράτη-μέλη τη Ένωση ε, έστειλαν διαστόματος των αρχικών και κυβερνήσεων και τη διακήρυξη ε, του Συμβουλίου ε, ένα χειρό μήνυμα για μια κοινή προσέγγιση για την προστασία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και θεσμών στην Ευρώπη. Σημειώνει το Συμβούλιο ότι το μίσος και ο αντισημιτισμός είναι ευρέως δεδομένο φαινόμενο ακόμη και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και για την μεγαλύτερη προστασία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Είναι ένα βασικό όχημα που επιτρέπει ε, την διάδοση της ρητορικής μίσους ε, για την καταπολέμηση της επιδημίας θα μπορούσε να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή ανταπόκριση και αντίδραση. Έχουμε συμπέρασματα Συμβουλίου για την εφαρμογή ε, του Χάρτη Μελλονδικαιωμάτων Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε τον ε, Οκτώβριο του 2017. Καλώ ορίζει τα μέτρα τη Κομισιόν και τη υψηλή ομάδας, της ομάδα υψηλού επίπεδου για την καταπολέμηση αρτισμού, αλλοδοξία και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης. Εμεί και υποστηρίζουμε τον συνεχιζόμενο διάλογο για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσου. Υπάρχει και ο κώδικας διοντολογίας που τροπολογήθηκε το 2016 από την Κομισιόν. Τέλος, θα πρέπει να θυμόμαστε και να εκφράζουμε την εκτίμησή μας για το σημαντικό έργο του Οργανισμού Θεμελιών Δικαιωμάτων. Ε, δεν έχουμε Μάλλον θα ήταν όλα αυτά τα μέτρα αναποτελεσματικά αν παραγνωρίζαμε το ρόλο της παιδείας ε, και της εκπαίδευσης των νέων. Θέλουμε τον εγγραμματισμό των μέσων, την κριτική σκέψη να προωθήσουμε ε, και να περιλάβουμε στην μαθησιακή διαδικασία και μεθόδους επίλυσης ε, κρίσεων και αντιπαραθέσεων. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση κλιμάτων μίσους μπορούν να ε, είναι αποτελεσματικά μόνο αν γίνεται καταγγελία από τα θύματα και αν δεν υπάρχει αστυνομική βία. Θα πρέπει επίσης αν έχουμε και τέτοια φαινόμενα να δηλώνονται ως εγκλήματα βίας. Πολλές φορές ε, όταν δηλώνονται, καταγγέλλονται τέτοιου είδους εγκλήματα από την αστυνομία δεν αναγνωρίζεται αυτό, αυτή η πράξη ως αξιόπινη. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα για την μετώπιση αυτού του προβλήματος. Θα πρέπει να δοθεί μεταξύ άλλων καθοδήγηση στους αστυνομικούς να συλλέγονται αναλυτικά δεδομένα για την αξιόπινη πράξη. Και επίση θα πρέπει να υπάρξει εργασία με την πεπειραμένη κοινωνία των πολιτών σε θέματα εγκλημάτων μίσου. Ε, εν συντομία, όλοι μα έχουμε ευθύνη. Πολιτική, εκπαιδευτική, κοινωνική λειτουργή, μαθητέ, φοιτητέ, γονεί και δικαστέ εισαγγελίε δεν θα πρέπει κανείς να κλείνει τα μάτια του ή τα αυτιά του και να υποκρίνεται ότι δεν βλέπει την αδικία αυτή, τη διακριτική μεταχείριση, το μίσος. Μετά το Άσβιτς έμαθε ο κόσμος ε, το μάθημά του και δημιούργησε ένα κόσμο που βασίζεται στην ειρήνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου. Είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Ευχαριστώ. Äh, σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αντιπρόεδρος, ε, κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, πριν από δύο εβδομάδε Είχαμε την επέτειο της 25 ης ε, την 25 η επέτειο την απελευθέρωση του Auschwitz Birkenau. Η Αριάννα Σέγκρε που επεβίωσε το ολοκαυτώματος μας είπε τη συγκινητική ιστορία της για τις απάνθρωπες βίες πράξεις ανθρωπότητες που αντιμετώπισε σαν μικρή κοπέλα. Μας υπενθύμησε ότι το μίσος, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός εξακολουθεί σήμερα να στοιχιώνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να θέτει σε κίνδυνο της, την ποικιλομορφία των κοινωνιών μας και τις μειονότητες που ζουν ανάμεσά μας. Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αποφύγει επανάληψη της ιστορίας και να διατηρήσει τις αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ένωση. Το ολοκαύτωμα μας έδειξε το ότι αντισημιτισμός και ο ρατσισμός που μπορούν να φτάσουν και η ανάμνηση αυτών είναι στο κέντρο του εγχειρήματο Ευρώπη, τη Ευρώπη, προστατεύει τι εβραϊκέ κοινότητε τη και όλε τι άλλε μειονότητε. Είδαμε ότι ο φόβο και το μίσο κατά του άλλου έχει γίνει κάτι κανονικό τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται κανονικό. Ανθεί στα βασικά μέσα ενημέρωση, στην πολιτική συζήτηση και στον κόσμο του διαδικτύου. Είναι σημαντικό πρόβλημα για όλη την κοινωνία μας και όχι μόνο για τις πληττόμενες ε, κοινότητες. Η αντισημιτική επίθεση κατά τη συναγωγή στο Χάλε είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα μόνο, αλλά καθημερινά οι μειονότητες γίνονται θύματα του μίσους στο διαδίκτυο και έξω το διαδίκτυο. Ήταν βασική η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίζει πρωτίστως την σωστή εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενσωμάτωση του Την οδηγία για την ισότητα την φιλητική ισότητα ε, και την απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τα κράτη-μέλη, με την κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ομάδα υψηλού επίπεδου κατά πολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για τα εγκλήματα μίσους και τους λόγους μίσους ε, στην ομοθεσία. Τα διάφορα σχετικά εργαλεία θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις πρακτικές ε, απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Συγκεκριμένες μορφές συνεδριάσεων της ομάδας υψηλού επίπεδου θα εξασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων από τα κράτη-μέλη να έχουμε απτά αποτελέσματα ανταποκρινόμενοι στις ομιλίες μίσους και στις πράξεις μίσους. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, ομιλίες μισαλλοδοξίας, πιέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για στεναρότερη δράση ξεκινήσαμε το δοντολογικό κώδικα για την καταπολέμηση παράνομων λόγω μίσου στο διαδίκτυο. Εκεί και διάφορες εταιρείε προσπαθούν, οι διάφορες πλατφόρμες εντός 24 ωρών έχουν προσχεθεί να εντοπίζουν και να κατεβάζουν ένα αναγκαίο το σχετικό περιεχόμενο. Έχει επιτευχθεί γρήγορη πρόοδος το 2016 μόνο 28% του περιεχομένου ε, το. Τώρα έχουμε ξεπεράσει το 70% και 89% των ε, διαφόρων ε, καταγγελιών εξετάζονται εντός του τακτικού προβλεπωμένου διαστήματος. Ε, Τον επόμενο μήνα θα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πέμπτης προσπάθειας εποπτείας μαζί με τις Κοινωνίε των πολιτών. Προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε όλους τους φορείς, κοινωνίε των πολιτών, τι εταιρείε του ίντερνετ και τι διάφορε αρμόδιε αρχέ για να ενισχύσουμε την ανταπόκρισή μα όσον αφορά του λόγου μίσου στο διαδίκτυο. Οι συντονιστέ μα για την καταπολέμηση ε, του, την καταπολέμηση του και του αντιμουσουλμισμού έχουν έρθει σε επαφή με τι διάφορε κοινότητε και ενίσχυσαν συνεργασίε και με του διεθνεί φορεί, με τα κράτη-μέλη, τις αρχές των κρατών μελών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης, εντατικά ε, προσπαθούμε να εφαρμοζώσουμε τη στρατηγική μας για τους Ρωμά και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις πράξεις κατά των Ρωμά. Η υιοθέτηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου για την καταπολέμηση αντισημιτισμού ήταν ακρογωνίως λήθος. Όλα τα κατημέλη ομόφωνα συμφώνησαν να επιδράσουν και προσεκλήθησαν να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές σχετικά με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε συγκεκριμένη ομάδα εργασίας να εξασφαλίσει συνέχεια στη δήλωση του Συμβουλίου και για να στηρίξει τα κατημέλη και τις ευρωπαϊκές κοινότητες ώστε να συνεργαστούν αναπτύσσοντας σχετικές στρατηγικές. Χαιρόμαστε που επερχόμενη Γερμανική Προεδρία ήδη ανακοίνωσε την πρόθεσή της την καταπολέμηση του αντισημιτισμού να τη βάλει πολύ ψηλά ως προτεραιότητα. Η στρέβλωση της κοινή μας ιστορίας ήταν ένα από τα βασικά σημάδια που τροφοδοτούσε τις φλόγες της διέρεσης και του μίσους, είτε γινόταν από τρίτες χώρες, είτε από τις ίδιες τις κοινωνίες μας. Σήμερα γίνονται προσπάθειες να παρνηθούμε, να στρεβλώσουμε τη μνήμη του ολοκαυτώματος, που καταπολεμούνται κάποιοι μόνο επειδή είναι Εβραίοι και εδώ αμφισβητείται η Ευρώπη. Προσπάθεια στρέβλωση τη ιστορία είναι κάτι που απειλεί τα θεμέλια μα. Η παραπληροφόρηση και οι ψευδεί ειδήσει επιτίθενται κατά του παρελθόντο, αλλά πρωτίστω επιτίθενται κατά του παρόντο μα. Οι δημοκρατίε μα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση και θα πρέπει να προσαρμοστούν δεόντω. πλατφόρμες στο διαδίκτυο έχουν χρησιμοποιηθεί για να δώσουν αυτά τα μηνύματα που χειραγωγούν την κοινή γνώμη και στρεβλώνουν τη δημοκρατική συζήτηση και παρεμβαίνουν στην πολιτική διαδικασία. Τέσσερις από, από τους πέντε Ευρωπαίους η παραπληροφόρηση είναι ένα πρόβλημα σε δημοκρατικό επίπεδο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η δημοκρατική η δημοκρατία προστατευμένη στην Ευρώπη. Για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη δημοκρατία μα και να την προστατεύσουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει σχετικό πρόγραμμα δράση τη δημοκρατία, θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση. Θέλουμε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση και θέλουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τι διαφημίσει τη πολιτικού περιεχομένου και να υπάρχουν καλύτεροι κανόνε για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία καθώ και ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε εξωτερικέ παρεμβάσει στα δημοκρατικά μα συστήματα από εκείνου που θέλουν να διχάσουν και να αποσταθεροποιήσουν την ένωσή μα. Αυτή είναι κοινή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τα κράτη-μέλη. Όπω το θεωρούμε το θέμα, οι μειονότητε δέχονται πιέσει και σήμερα και γι' αυτό θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ζουν τη ζωή τους ελεύθεροι χωρίς να έχουν την απειλή του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και του σχετικού μίσους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την ε, ομάδα τη διακομματική κατά του ρατσισμού και για την ποικιλομορφία και την ομάδα εργασίας για τον αντισημιτισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων. Πρώτη η κυρία Μέτσολα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα πολλές ομιλίες, αλλά αυτή που δεν θα ξεχάσω ήταν του Μαριον Κιούρσκι που κατάφερε να βγει από το Auschwitz. Και είπε ότι η διαφορία πρέπει να σταματήσει, ότι το Auschwitz δεν μας ήρθε από τον ουρανό, έγινε σιγά σιγά, γιατί πάρα πολλοί έκλειναν τα μάτια και δεν φρόντιζαν για δικαιοσύνη. Πολλοί βρίσκαν από διοπαμπέους τράγου και πολλοί δέχτηκαν ότι δεν θα έπρεπε να έχουν δεχτεί. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τον ασημιτισμό, τον ρατσισμό και το μίσο στην κάθε του έκφραση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πάρα πολύ καλά την φρίκη και πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Πρέπει λοιπόν να διδάσκουμε τον κόσμο όχι μόνο για το τι συνέβη, αλλά και για το πώς συνέβη, σιγά, σταδιακά. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να μάθουμε τα μαθήματα της ιστορίας και το όταν δεν θα υπάρχουν πια επιζήσοντες για να τους ακούμε. Οι επιθέσεις που γίνονται κατά των Εβραίων ή συναγωγών βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν από δύο Πομπέι τράγοι και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι πολύ αργά προχωράμε για να υποστηρίξουμε τις αξίες μας. Απειλούνται οι αξίες μας σε πολλά σημεία της Ευρώπης. Δεν μπορούμε λοιπόν να σιωπούμε όταν οι Ευρωπαίοι ζουν με μια βαλίτσα δίπλα στην εξώπορτα, μπας και πρέπει να φύγουν. Πρέπει να αγωνιζόμαστε για τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και να μην βρίσκουμε άλοθη. Η ευρωπαϊκή μας ιστορία πολύ συχνά χτίστηκε σε βάρος των έφραστων. Όταν λέμε ποτέ ξανά να το εννοούμε και αυτό σημαίνει να αναλαμβάνουμε δράση. Να μην ξεχνάμε την ε, δέκατη εντολή που λέει ότι δεν πρέπει να διαφορούμε για τον πλησίον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πύρη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πριν από 75 χρόνια, εμείς οι Ευρωπαίοι συμφωνήσαμε ποτέ ξανά. Κι όμως το 2020 εξακολουθεί να υπάρχει άνοδος του αντισημιτισμού, να υπάρχει μυσαλλοδοξία. Τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και εδώ, δημιουργούν ένα κύμα ρατσισμού με τη ρητορική τους κατά της ε, είτε πρόκειται για τους Ρώμα, είτε πρόκειται για ε, τους Εβραίους, είτε και οποιοδήποτε άλλον. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ρητορική ε, των λαϊκιστών. Δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει μια κοινή μας πολιτική, να αποτελέσει μια κανονικότητα. Όχι, ούτε μπορούμε να δεχτούμε ε, τρίτες πλευρές όπως είναι το FDA στη Γερμανία, το FIDE στην Ουγγαρία, είτε άλλοι στην Ιταλία κλπ. να κυριαρχήσουν ε, εδώ. Όχι, εμείς πάντα θα είμαστε υπέρ της ελευθερίας, ελευθερίας για όλους, για ό,τι θέλεις να είσαι, για να πιστεύεις ό,τι θέλεις να πιστεύεις. Πρέπει να δεσμευτούμε πιο έντονα κατά ε, της ρητορικής μίσους. Θα, θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε υπέρ των μειονοτήτων, των ευάλωτων και να τους προστατεύουμε από παντός είδους διάκριση. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να σέβεται το δίκαιο και όχι το δίκαιο έτσι γενικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν να θυμόμαστε αυτά τα 75 χρόνια που πέρασαν από την ε, έξοδο από το Auschwitz. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δρούμε κάθε φορά που υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος κάποιων. Ευχαριστώ κυρία Φρεντερικ Ρίς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 37 χρονών θα ήταν α, ο ένας, ένας οποίος ε, πριν από 14 χρόνια ε, δολοφονήθηκε σε εργατικές κατοικίες ε, στο Παρίσι, άρα λιμή συγκεκριμένα. Και μάλλον επειδή ήταν Εβραία, την πέταξαν και από το παράθυρο δεν θα δικαστεί όμως ο δράτης. Θεωρήθηκε ότι δεν ε, ήταν ε, σε ε, κατάσταση λογική γιατί ήταν υπό την επίρρεια της κάναβης. Έχουμε λοιπόν φαινόμενα αντισημιτισμού που σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους που σήμερα, ακόμα και σήμερα επειδή είναι Εβραίοι, Πρέπει να προστατεύσουμε κημητήρια, σχολεία και άλλα ε, εβραϊκά κτίρια. Πρέπει να θυμόμαστε το ολοκαύτωμα, να θυμόμαστε και να εκπαιδεύουμε. Όταν όμως έχουμε ρατσιστική βία που μαστίζει πόλεις σε κοινωνικά δίκτυα, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν πρέπει να το ανεχόμαστε. Πρέπει να το καταδικάζουμε, να το τιμωρούμε. 50 και κρατών και κυβέρνηση πήγαν στην Ιερουσαλήμ για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Auschwitz. Και ο πρόεδρος Ούγκρου ήταν εκεί, της ήταν εκεί και είπε και στη Βουδαπέστη παρόλα αυτά Χιλιάδες Ναζί συγκεντρώθηκαν από τέσσερις γονείς του κόσμου για να παρελάσουν για την ημέρα τιμής, ε, για να τιμήσουν ε, τους ήρωες του Τρίτου Ράιχ. Αν είναι δυνατόν, ε, πώς μπορούμε να πούμε ότι κάνει αρκετά Ευρώπη σήμερα. Mm. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίλιπ Ντεμάν. Αγαπητοί συνάδελφοι, Μιλάμε για τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. Η συζήτηση αυτή γίνεται και στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Παντού υπάρχουν και ναζί και ρατσιστές και αντισημιτιστές, αλλά το πραγματικό πρόβλημα δεν το κατονομιάζουμε συνήθως. Το ρεύμα που υπάρχει από μουσουλμάνους ρατσιστές οι οποίοι είναι υπέρ κατά το 99% του αντισημιτισμού στην Ευρώπη. Ποτέ δεν το λέμε αυτό. Μιλάμε για τους Ναζί, αλλά τελικά εσείς είσαστε μακριά από την πραγματικότητα. Ονομάστε τους εθνικιστές ρατσιστές, επειδή θέλουν να προστατεύσουν τα δικά μας τα σύνορα. Λύση υπάρχει για τα προβλήματα. Και η λύση σίγουρα δεν είναι αυτό που προτείνεται. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαστε κάπως πιεσμένοι από πλευράς χρόνου. Γι' αυτό θέλω να σας πω εκ των προτέρων ότι μόνο πέντε συνάδελφοι θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Επόμενος, ο κύριος Λαγκοντίνσκι, ο Σεργέη. Mm. πολύ ε, όταν είδαμε τι γίνεται με τους ακροδεξιούς τους φίλους αυτού που μόλις πριν πήρε το λόγο ε, εξέλεξαν τον Τόμας ε, και Μεριχέ στην Θουριγγία. Βλέπουμε να χρησιμοποιούνται αντισημιτικά κλισέ και όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Αυστρία, στη Λετωνία. Ενώ Εβραίοι εδώ στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι, οι Εβραίοι, οι που δεν νιώθουν καλά και πραγματικά θα πρέπει να πάψουν ε, να ισχύουν, θα πρέπει να καταρρεύσουν αυτές ε, οι, ε, οι προκαταλήψεις και αυτά τα στερεότυπα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να γίνονται εγκλήματα που έχουν αντιεβραϊκά κίνητρα. Θα πρέπει λοιπόν να σπάσουμε τα φράγματα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και Στρέφομαι σε όλους μας, ε, στα κράτη-μέλη, στην Κομισιόν. Καλές, ε, καλά λόγια στην Ιερουσαλήμ από την Πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν φτάνουν όμως αυτά. Χρειαζόμαστε να σπάσουμε αυτά τα φράγματα. Χρειαζόμαστε δράση πραγματική. Τι θα κάνουμε ε, έχουμε την, ε, την απεσταλμένη κατά του αντισημιτισμού, την αντιπρόσωπο. Έχει επαρκή εντολή, μπορεί να κάνει πραγματικά αυτό που πρέπει. Πώς θα τα εφαρμόσουμε στην πράξη, τι πιστεύετε. Δεν έχουμε απαντήσεις και αυτές τις απαντήσεις ε, περιμένουμε. Και δεν τις περιμένω μόνο ως μέλος της ομάδας εργασίας κατά του αντισημιτισμού. Το χρήση πρέπει λοιπόν να κρατήσει κρατήσουμε ε, τη, τη στάση αυτή που πρέπει. Ευχαριστώ. δόλο ολοκληρώνω τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς άλλος να πάρει το λόγο πέραν των έξι που έχω καταγράψει μέχρι τώρα. Άρα σταματά εδώ και επόμενος ε, ο κύριος Προκατσί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αρκούσε να είναι κανείς αυτή την αίθουσα εδώ και δύο ώρες για να ακούσει λόγια μίσους και αντισημιτισμού. Δύο ώρες πριν, ο λαός του Ισραήλ κατηγορήθηκε για απατχάιτ, για εκμετάλλευση των Παλαιστινίων, ε, βία προσάρτηση, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εγκλήματα πολέμου, το να λέμε αυτά τα πράγματα, ήταν οι ίδιοι που κρύβονται από την ευθύνη για το ριζοσπαστικό Ισλαμισμό. Πίσω από εκεί για τις επιθέσεις αντισημιτικές στην Ευρώπη. Οι ίδιοι είναι όσον αφορά στον ευρωπαϊκό λαό να μπορεί να ασκήσει τις δικές του θρησκευτικέ παραδόσεις στην Ευρώπη και ίσως έχει δίκιο ο Goldsmith, ο πρόεδρος της διάσκεψης των ραβίνων, των Ευρωπαίων ραβίνων, που πριν από μερικές εβδομάδες στην Ιταλία είπε σήμερα τα περισσότερα προβλήματα τα έχουμε από την αριστερά. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία όσον αφορά το μέτωπο του αντισημιτισμού. Η κυρία Ernst έχει τώρα το λόγο. είπε κάποια πράγματα ο ε, προλαλής και στράφηκε κατά της αριστεράς. Ε, πράγματι έχουμε συναγωγές που γίνονται θύμα ακροδεξιών αλλά υπάρχουν ένοπλοι ε, οποίοι θα πρέπει να τα φυλάσουν αυτά τα κτίρια ε, και πραγματικά υπάρχουν πολλοί Εβραίοι οι οποίοι νιώθουν ότι κινδυνεύουν. Ο αντισημιτισμός περιγράφεται στην ιστορία με τελείως διαφορετικά λόγια από ό,τι θα έπρεπε και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε και το σωστό, τα σωστά λόγια να χρησιμοποιήσουμε με λόγια και με πνεύμα να στραφούμε κατά των ναζιστών στην κοινωνία, στο δρόμο, στην πόλη, μέσω της δικαιοσύνης, ε, στο κοινοβούλιο, στην καθημερινότητα και επίσης ε, θα πρέπει ξεκάθαρα να καταδικάσουμε δεν ήταν το ίδιο φασισμός ε, και και ο κομμουνισμός γιατί και εδώ δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όπως πρέπει. Σίγουρα υπάρχουν θύματα του φασισμού και του ρατσισμού και τους χρωστάμε και στους δύο. Ευχαριστώ. Κυρία Φεράρα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαινόμενα όπως ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ε, ομοφοβία και άλλες μορφές μη ε, χτυπάνε συναγερμό σε πολλα κάτι κράτη-μέλη δημιουργούν μίσους και προκατάληψη ή έχουν διάδοση ανησυχητική και στο διαδίκτυο και εκτός αυτού. Να προστατεύονται κοινωνικές ομάδες και άνθρωποι οποιοδήποτε μορφή διάκρισης και βίας για λόγους που συνδέονται με το χρώμα της επιδερμίας, τη θρησκεία, τις προσωπικές απόψεις ή το σεξουαλικό προσανατολισμό σημαίνει όχι μόνο να εγγυόμεθα σε όλου την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και να έχουμε μια κοινωνία που θα είναι πιο συνεκτική και θα καλύπτει του πάντε. Χρειάζεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να θετήσουν πρωτοβουλίε και μέτρα πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, κυρίω για του πιο νέου, όσον αφορά τα εγκλήματα και τι διάφορε ομιλίε μίσου, παρακινού στο μίσο. Δεν, δεν γίνεται επαρκή δίωξη και καταγγελία παραμένουν ατιμόρυτε πράξει και αυτό έχει μεγάλη συνέπεια όσον αφορά την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων. Και για το κοινό όφελο τη Ευρώπη πρέπει να αντιστραφεί αυτή η τάση που διαπιστώνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πόλακ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι πιστός και πολλοί από εσάς φαντάζομαι ότι πιστεύετε Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι, δείχνουν συμπάθεια στους ε, φασίστες ε, και παρουσιάζονται ως ε, πιστοί. Όμως ε, βλέπουμε ε, να είναι δυνατή μια νεοναζιστική κυβέρνηση. Εκεί πια ε, πρέπει να χτυπάει το καμπανάκι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε όταν όλοι έχουμε το ίδιο αίμα και να λέμε για το διαφορετικό χρώμα δέρματος ή τα κτλ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μάλλον δεν υπάρχει διάκριση. Το ίδιο αίμα τρέχει στις λέβες ε, όλων. Οι φασίστες πραγματικά έκαναν ε, αποτροπιαστικές ε, πράξεις και λέγαν ότι αυτά το έκαναν, τα έκαναν στο όνομα του Θεού και του λαού. Έτσι αιτιολογούσαν τις πράξεις τους. Επίσης, έχουμε φτωχές περιοχές με άτομα που ζουν σε συνθήκες φρικτές, δεν έχουν απογέτευση, δεν έχουν πόσιμο νερό ε, ε, και αν αγνοήσουμε αυτά τα προβλήματα, τότε θα ε, εκμεταλλευτούν οι φασίστες και πρέπει να πω ότι οι πολιτικοί πρέπει να ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα και θα πρέπει να αποφύγουμε να μας ξεπεράσουν τα πράγματα, όλες αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να τις χαρακτηρίζουμε εγκλήματα, παραπτώματα και θα πρέπει έτσι να δράσουμε. Όλοι γνωρίζουμε ποιος, ε, πού οδηγεί ο εξτρεμισμός. Αν του δώσουμε την ευκαιρία του εξτρεμισμού, ξέρουμε πού θα καταλήξει, ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σε πολλά χρόνια οι ε, εξτρεμιστές βασίζονται στη διαφθορά, στα τα προβλήματα ε, και καταγγέλνουν τους Ρωμά. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να ανταλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί μαστίζουν την Ευρώπη πραγματικά. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ο κ. θα Αγγιλάρη, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε Γιούροβα, η συζήτηση αυτή κατά του αντισημιτισμού και του ρατσισμού αλλά και του μίσου στην Ευρώπη έχει πολύ νόημα και είναι και φορτισμένη. Όχι γιατί το ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι αυξάνονται οι δράσεις διακρίσεων σε βάρος κάποιων ανθρώπων ή κατηγοριών ολόκληρων ε, Ευρωπαίων πολιτών, των οποίων τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και γιατί αυξάνονται ε, τα εγκλήματα μίσου και η ρητορική μίσου σε βάρο αυτών των ανθρώπων και αυτών των κατηγοριών. Εξού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χρέο να εκφράσει την ανησυχία του, αλλά να δείξει ότι είναι διατεθειμένο να αντιδράσει. Και το Συμβούλιο επίσης να δώσει αυτή τη μάχη και να ενισχύσει ό,τι εργαλεία διαθέτουμε στη διάθεσή μας. Από τον Ιούνιο του 2017 έχουμε το ψηφισμά μας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και έχουμε δείξει ότι δεν θέλουμε να υπάρχει αρνητισμός απέναντι στο ολοκαύτωμα. Αλλά περιμένουμε και από το Συμβούλιο. Το Δεκέμβριο του 2018 ζητήσαμε πάλι τα εργαλεία, την εκπαίδευση κατά του μίσους, αλλά και τις κυρώσεις κατά των εγκλημάτων μίσους, που οδηγούν στη βία. Πρέπει λοιπόν αυτή η απόφαση πλέον το 2018 να τεθεί σε εφαρμογή υπάρχει στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Πρώτον, κατάρτιση των αρμοδίων αρχών. Δεύτερον, μητρό για τις περιπτώσεις αυτές μίσους. Και τρίτον, προστασία των θυμάτων και εγγυήσει απέναντι σε αυτούς που απειλούνται όχι μόνο ε, για τους Εβραίους, αλλά εδώ πέρα πρόκειται και για τους Αθήκανους, αλλά και για άλλους που είναι θύματα ρητορικής μίσους και δράσεων μη δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιες δράσεις γιατί βρίσκονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Γιούλια Ντόνατ. Ευχαριστώ πολύ. Στην Ουγγαρία τελευταία μια εκστρατεία της κυβέρνησης κατά τον Ρώμα υπήρξε και τα έβαλε με τα παιδιά των Ρώμα στην Ήπεθρο. Επρόκειτο για τα επιδόματα που έπαιρναν τα παιδιά αυτά και κάποιοι τα έβαλαν μαζί τους λέγοντας ότι παίρνουν τα επιδόματα αυτά χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Όντως η ρητορική μίσους αυξάνεται σε πολλές χώρες μας. Τα τελευταία χρόνια αντί να περιορίζεται, αντίθετα ενισχύεται ακόμα περισσότερο δημιουργούνται πάλι από διοπομπέοι τράγοι και φόβος επειδή αλλάζει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να δράσουμε τώρα γιατί αλλιώ θα έχουμε ένα ντόμινο. Πρέπει να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Για παράδειγμα, οι πρακτικές νομοθεσίας με αποκλεισμούς, η προπαγάνδα γενικότερα. Πρέπει να δράσουμε τώρα για τελειώς υπονομεύουμε τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η αλληλεγγύη, η ανθρώπινη εξωπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η μη διάκριση. Χωρίς αυτά δεν θα έχουμε ρόλο να παίξουμε στο μέλλον. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Η Σουζάνα Τσεκάρντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ιστορία του δυτικού κόσμου απέδειξε ότι ε, δείχνει την, ε, ε, το πώς καταραίει τελικά μια κοινωνία. Λοιπόν, όποιο βλέπει να δεν θέλει να καταραίει η κοινωνία, πρέπει να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό. Η καταπολέμηση πρέπει να προβλέπει την, την προστασία του ειδευτικού ακαιρεότητα του Ισραήλ, την πολιτική και θρησκευτική. Διότι το Ισραήλ είναι στην πρώτη γραμμή τη δημοκρατική ελευθερία στη Μέση Ανατολή η συνεισφορά που η χριστιανική παράδοση έδωσε στη διαμόρφωση της δυτικής ε, κοινωνίας και του πολιτισμού ήταν θεμελιώδη σημασία. Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού σημαίνει όχι μόνο να υπερασπιστούμε το Ισραήλ που ταυτόχρονα είναι η πατρίδα του Εβραϊσμού και προστατεύει την μνήμη του χριστιανισμού, αλλά να προσπιστούμε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ισλαμική τρομοκρατία, από τον φονταμεταλισμό, το σκεφτικό και κάθε κίνημα κατά της ελευθερίας και κατά της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε. κυρία Κούνκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. σχεδόν, ε, σχεδόν λέω, είναι πειρασμός ε, να ακούμε ωραία λόγια ότι αγωνιζόμαστε ε, για να αντιμετωπίσουμε ε, τη, τη και το ρατσισμό. Είναι κενά λόγια, το γνωρίζουμε ε, σε πολλές περιπτώσεις. Πίσω από τη ρητορία αυτή υπάρχουν όμως από πίσω άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που δεν τα λαμβάνουμε υπόψη το όνομα που έχει κάποιος, ποιοι είναι του, ε, το υπόβαθρό του, όλα αυτά ε, οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση και πραγματικά εξαπλώνονται σαν τη φλόγα και πρέπει να τα πάρουμε πολύ σοβαρά. Πρόκειται για απειλέ ε, πάρα πολύ σοβαρές. Είναι απαράδεκτο η αρχική κρατού και κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκής Ένωση να μην καταφέρουν μέσα σε 15 χρόνια να υπογράψουν την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Είναι αλήθεια ότι η συζήτηση για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια. Αν συζητάμε για αλήθεια, ε, δεν πρόκειται για ε, να ζει ή 75 χρόνια μετά την απελευθέρωση του Auschwitz πρόκειται για την απελευθέρωση του ναζιστικού στρατοπέδου στο Auschwitz. Εμένα με εξέπληξε όταν οι αριστεροί διαφωνούν με ε, αυτά που εμεί θέλαμε και ψηφίσαμε για τον κομμουνισμό. Να θυμίσω ότι είχε πει ο Στάλιν που είχε πει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να βγάζουν το θυμό τους απέναντι στους Εβραίους όταν θα τελειώνουν την εργασία τους. Και στον πολωνικό στρατό είδαμε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα θυμίσω ότι είπε η Πολυνόφσκα που είναι συγγραφέας από την Πολωνία. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και δεν μπορούμε να αρνούμεθα το τι πραγματικά συνέβη. Ε... Πονσάτιο Μπιόλς. Ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα χειρότερα εγκλήματα κατά των Εβραίων έλαβε χώρα το 1492 όταν οι καθολικοί βασιλείς έδιωξαν ε, τους Σεφαρδίτες. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο αντισημιτισμού από πλευράς του κράτους. Κάτι που θαύμασε ο Αδόλφος Χίτλερ και προσπάθησε να το επαναλάβει και αποτελεί ακρογωνίο λίθο του τραγικού μητρώου που έχει η Ισπανία όσον αφορά τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό. Τώρα το βλέπουμε και σε βάρος της καταλωνικής μειονότητας. Το Ίδρυμα Φρανσίσκο Φράγκο, για παράδειγμα, παραμένει νόμιμο και οι Ισπανοί δικαστές χρησιμοποιούν ε, νόμους σε βάρος των ε, Καταλανών. Εμείς δεν ζητάμε προστασία των ε, μειονοτήτων από τριτορική μίσου, ζητάμε όμως δικαστές οι οποίοι να μην προωθούν τέτοιες διακρίσεις. Ευχαριστούμε συνάδελφος Στομπέ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι.